Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών, ιδιαίτερα την αυτού εξοχότητα πρέσβη του Ελ Σαλβαδόρ, την κυρία Βιλατόρο, την αυτού εξοχότητα πρέσβη της Νικαράγουα, τον κύριο Μόντες, να καλωσορίσω τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Αφέλτ, προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στη Διεύθυνση για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική, την κυρία Φερνάντε Ντελαπουέντε, υπεύθυνο του τμήματο εκλογική παρατήρηση Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και να σα πω ότι η διερμηνία παρέχεται στη, στα αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά και παθητικά στα γαλλικά. Το σχέδιο τη ημερήσια διάταξη έχει διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν στα αγγλικά, ελληνικά και στα ισπανικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα θεωρηθεί ότι συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο σημείο, στις ανακοινώσεις, κύριοι συνάδελφοι. Στις 31 Αυγούστου του 2018, η κυβέρνηση της Γουατεμάλα αποφάσισε να μην ανανεώσει την εντολή της ΙΣΥΚ της Διεθνούς Επιτροπής κατά της ατιμορρησίας στη Γουατεμάλα μετά το 2019. Θέλω να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό και τη λύπη μου για την απόφαση αυτή, η οποία συνιστά ξεκάθαρη οπισθοδρόμηση στην εδραίωση και διασφάλιση του κράτους δικαίου. Όπω γνωρίζετε, η συσήξη στάθηκε κατόπιν αιτήματο της κυβέρνηση της Γουατεμάλα και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη συνεχιζόμενη διαδικασία προώθησης των μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση των κρατικών θεσμών, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην καταπολέμηση τη ατιμορρησία με την αποκάλυψη πολυάριθμων σκαδάλων διαφθοράς. Από το 2007 μέχρι και σήμερα, η ΣΥΣΥΚ έχει διενεργήσει περισσότερε από 200 έρευνε εκ των οποίων οι περισσότερες, περισσότερες από τις 160 έχουν οδηγήσει σε απαγγελίες κατηγοριών εναντίον προέδρων, υπουργών, πρώην διευθυντών της Εθνικής Αστυνομίας, απόστρατων στρατηγών, πολιτικών, επιχειρηματιών, εμπόρων ναρκωτικών, εκτελεστών κτλ. Κύριοι συνάδελφοι, όπω γνωρίζετε, η αντιπροσωπεία μα έχει επανειλημμένα στηρίξει το έργο και την εντολή τη ΣΥΣΥΚ. Για τον λόγο αυτό, σα θυμίζω ότι το Προεδρείο τη Αντιπροσωπείας για τι σχέσει με τι χώρε Κεντρική Αμερική εξέδωσε πριν από λίγου μήνε δήλωση που την υπέγραψα εγώ με την ιδιότητα τη Προέδρου και του δύο αντιπροέδρου σχετικά με την απέλευση του Επιτρόπου Μπελάσκεθ από την Γουατεμάλα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή μα επισκέφθηκε τη Γουατεμάλα από τι 16 μέχρι τι 18 Φεβρουαρίου του 2015 και ότι με την ευκαιρία αυτή είχε μια μακριά και ενδιαφέρουσα συνάντηση με αντιπροσώπου τη ΕΣΥΚ και με τη Γενική Εισαγγελέα τη χώρα, κυρία Αλντάνα, και η γενική εκτίμηση που αποκομίσαμε σαν αντιπροσωπεία είναι ότι επιτελεί ουσιαστικό και σημαντικό έργο και προσδοκούμε τουλάχιστον ότι η κυβέρνηση θα της επιτρέψει να συνεχίσει απρόσκοπτα το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει μέχρι τη λήξη της εντολής της. Η ΣΥΣΥΚΑ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τη Γουατεμάλα στην ίσχυση του κράτους δικαίου και της θεσμικής ικανότητας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, αλλά και πέρα από την ημερομηνία αυτή, πάντα προ όφελο όλων των πολιτών τη Γουατεμάλα στο σημείο 3 που αφορά στην έκθεση της αποστολής των εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κοινοβουλευτικές και δημοτικές εκλογές στο Ελ που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαρτίου του 2018. Όπως γνωρίζετε, στις 4 Μαρτίου διεξήχθησαν στο Ελ Σαλβαδόρ βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη 84 μελών της νομοθετικής συνέλευσης και 262 δημάρχων. Κατόπιν πρόσκληση τη κυβέρνηση του Ελσαλβαδόρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε αποστολή εκλογικών παρατηρητών στη χώρα με επικεφαλή στον Ευρωβουλευτή κ. Ιντρουκουάιθ και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσε σαν επικεφαλή στον Ευρωβουλευτή κύριο Λοπέ. Η αποστολή των εκλογικών παρατηρητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την τελική έκθεση τη αποστολή στι 22 Μαου του 2018 στο Σαν Σαλβαδόρ. Έπειτα από δύο αναβολέ τη παρουσίαση τη έκθεση σε αυτή την αντιπροσωπεία, θα έχουμε επιτέλου την ευκαιρία να ακούσουμε τα ευρήματα τη αποστολή των εκλογικών παρατηρητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Ιντουρκάιθ, επικεφαλή τη Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών στο Ελ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σε όλου, Κύριε και κύριοι. Σε αυτή την ε, παρουσίαση τη εκλογική, της αποστολής για την ε, παρατήρηση των εκλογών, ε, ναι, στο Σαλβαδό στις 4 Μαρτίου του 2018 για τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Επιτρέψτε μου τα πρώτα μου λόγια να είναι λόγια ευχαριστειών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που πλαισίωσαν τον επικεφαλής και κατέστησαν αυτή την ε, Επιτροπή για την Προσωπή Εκλογικής Παρατήρησης μια επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μιλώ για τους εκπροσώπους ε, Τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και ιδιαίτερα την κυρία Κόντσα Φερνάνδεθ Ντελαπουέρτε που μα συνοδεύει, και παρίσταται. Επίση, μια ομάδα που είχε πάει πριν από εβδομάδε και μήνε ολόκληρου, υπό την ηγεσία του Αλεξάνδρ Γκρέι. Καλά, δεν θα αναφέρω τώρα όλου όσοι συνεισέφεραν, αλλά ξέρουν ποιοι είναι. Ήταν πραγματική κινητήρια δύναμη για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η αποστολή μας. Τούτων ορών λεχθέντων, Θέλω να τονίσω και τη δουλειά που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και όλοι οι βουλευτές που πήγαν στο Σαλβαδόρ. Ο Χαβι Λόπεθ ε, ήταν επικεφαλής, σοσιαλιστής, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ε, πραγματικά συνεργαστήκαμε πάρα πολύ αγαστά στο Σαλβαδόρ. Τώρα, για να μπούμε στην ουσία, κυρία Πρόεδρε, με την άδειά σα, ε, τι έγινε στις εκλογές. Θα ήθελα να βάλω έτσι μια επικεφαλίδα, ένα τίτλο, αν θέλετε, για το τι συνέβη εκεί. Πώς θα το χαρακτήριζα. Ήταν υπόδειγμα οι εκλογές αυτές, παράδειγμα προσμίμηση μίμηση για την Κεντρική Αμερική, αλλά και για τον κόσμο όλο. Πραγματικά, θυμάστε τι είχε γίνει άλλες φορές σε προηγούμενες εκλογές στο Σαλβαδόρ και γνωρίζοντας και γενικότερα το κλίμα που επικρατούσε στην περιοχή, στο παρελθόν, στη Γουατεμάλα, είδαμε τι συνέβη στην Ιγαράγουα, στην Ονδούρα. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι το Σαλβαδόρ έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη. Ήταν οι εκλογές ε, πάρα πολύ καθαρές, ε, πάρα πολύ γνήσιες, ε, με μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα και την, ε, το εκλογικό δικείο. Και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι όλοι θυμόμασταν τι είχε γίνει το 2015 και η σύγκριση με τη φετινή χρονιά ήταν πολύ εύγλωτη. Πολύ καλύτερες εκλογές, πρόκληση ήταν αυτή πραγματικά πολύ δύσκολη ε, και περίπλοκη γιατί το εκλογικό σύστημα, ξέρετε, και θα πω δύο λόγια στη συνέχεια γι' αυτό, είναι περίπλοκο, πάρα πολύ δύσκολο για τις βουλευτικές εκλογές. και είναι δύσκολη στη διεξαγωγή τους η εκλογική και η αναμέτρηση. Από τα ψηφοδέλτια τα ίδια δηλαδή μέχρι την όλη διοργάνωση νομίζω πήγανε πολύ καλά και βελτιώθηκε πολύ η διαδικασία σε σχέση με την εκλογική αναμέρτηση του 2015. Υπήρχαν όλα τα εκλογικά τμήματα και η διαβίβαση των αποτελεσμάτων ε, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, γιατί αμφέβαλαν πώς θα γινόταν η μετάδοσή τους κτλ. Ωραία. Ε, ποιο είναι τώρα το καινούριο και το θετικό, αν μου επιτρέπετε, στις εκλογές αυτές. Δεν ήταν τόσο πολύ κομματικά φορτισμένες, γιατί συμμετείχαν περισσότερο οι πολίτες ε, στις εκλογές και λιγότερο τα κόμματα. Αυτή η συμμετοχή των πολιτών συνοδευόταν και από μια χειραφέτηση των πολιτών δηλαδή που συμμετείχαν ενεργά στα εκλογικά τμήματα. Και αυτό ήταν χάρη στο ανώτατο εκλογοδικείο που είχε δύσκολο ρόλο με τα όσα είχαν ζήσει στο παρελθόν, τις προηγούμενες εκλογές και τους προηγούμενους μήνες. είχαν κάνει κάποιες δοκιμές και με μεγάλη δυσκολία, αλλά τελικά πραγματικά πήγαν πάρα πολύ καλά, τέλεια. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω για τα σταλίες και παρατυπίες, γιατί όταν ακούσα τα σταλίες, ο κόσμος ε, νομίζει ότι υπήρχε καμία μεγάλη νοθεία στις εκλογές ή τεράστια προβλήματα. Θα έλεγα ότι υπήρξαν κάποιες αδυναμίες στη διαδικασία, αδυναμίες. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν θα το έβγαζα σε εφημερίδε και στι δικές μας χώρες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, Κάποιε αδυναμίες στα εκλογικά τμήματα όταν έχουμε εκλογέ. Ποια ήταν αυτά τα ασθενή λοιπόν σημεία, τα οποία και αυτά τα σημειώσαμε στις συστάσεις που κάνουμε. Η ομάδα παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να προσθέσω και το εξής. η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήμασταν εμείς, ήταν εκείνοι που ήταν παρόντες σε όλη τη χώρα, σε όλα τα διαμερίσματα. Έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπήρξε διαμέρισμα που να μην είχε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε στο Σαν Σαλβαδόρ, που είναι η πρωτεύουσα, είναι προφανές να υπάρχει τέτοια παρουσία, αλλά υπήρχε και εκεί που είναι πιο κατοικημένε περιοχές της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά κυριάρχησε με την παρουσία της. Ποιε ήταν οι αδυναμίες λοιπόν ε, που σημειώσαμε και το έχουμε βάλει και στα συμπεράσματα, όπως είπα και προηγουμένω, και στι συστάσεις μα. και το δώσαμε και στην κυβέρνηση και στα κόμματα και στο εκλογοδικείο σε μετέπειτα επίσκεψη μετά τις εκλογές. Λοιπόν, ήταν αυτές οι δυναμίες. Υπήρχε μια δυσκολία στο μητρό των υποψηφίων, στην καταχώρησή τους, γιατί το ανώτατο εκλογοδικείο είχε προβλήματα, δεν μπορούσε να ε, διασταυρώσει τα στοιχεία και ε, τα έγγραφα των υποψηφίων. Το διαπιστώσαμε και εμείς αυτό δεν είχε αρκετό προσωπικό ή αρκετούς πόρους. Επίσης, το εκλογοδικείο που μας το είπαν εκεί οι ίδιοι, δεν μπόρεσε να διερευνήσει κάποιες παραβιάσεις που έγιναν και παρατυπίες σε εκλογικά τμήματα. Αυτό έχει να κάνει με την ίδια την εκλογική διαδικασία και πώς εκτελείται ο εκλογικός νόμος. ήταν δεμένα ε, και τα χέρια του δικαστηρίου και τα, τα πόδια του. Ε, δεν, είχαν μεγάλη δυσκολία ως προς τη διασταύρωση των εγγράφων. Και κάτι άλλο, το ίδιο το δικαστήριο δεν μπόρεσε να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών κομμάτων όχι, διορθώνει ο μιλητή, όχι να χρηματοδοτήσει το ίδιο, να ε, εξακριβώσει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, από πού προέρχονται τα χρήματα. Για, γιατί ο νόμος δεν επιτρέπει στο εκλογοδικείο να αναμειχθεί σε τέτοια θέματα. Αυτά σε ό,τι αφορά το ε, εκλογοδικείο. Αυτές ήταν κάποιες αδυναμίες, αλλά όχι παρατυπίες ή ατασταλείς. Ένα δεύτερο θέμα ε, που προερχονται τα χρηματα γιατι ο ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ή κάποια σφάλματα ε, ήταν εκλογικοί κατάλογοι αυτοί καθ' αυτή. Ε, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ε, πολλές φορές στις λατινοαμερικανικές χώρες ε, συμβαίνει υπερβολικά συχνά. Ε, στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται νεκροί που δεν τους έχουν διαγράψει ή κρατούμενοι τους οποίους τους έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα ή πολλοί ε, μετανάστες που έχουν αποδημήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπάρχει μεγάλη διασπορά από το Σαλβαδόρ, ε, άνθρωποι που ζουν στις Ηνωμένε Πολιτείες και αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς κατάλογους και δεν τους διαγράφουν από εκεί. Λοιπόν, χρειάζεται ε, ενημέρωση των καταλόγων και ε, έτσι κάπως να, να καθαρίσουν λίγο οι εκλογικοί κατάλογοι. Ένα άλλο σημείο την ημέρα των εκλογών δεν γίνεται ε, σεβαστή η περίοδος περισυλλογής ε, που επιβάλλεται από τον νόμο, την παραμονή και την ίδια ημέρα των εκλογών. Το ξέρει αυτό η πρέσβης. Το έχουμε πει παντού ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα ενός πολιτικού κόμματος. Δεν σέβονται αυτή την περίοδο. Συνεχίζουν την προεκλογική εκστρατεία, την προπαγάνδα, τα κόμματα μέχρι το εκλογικό τμήμα με μπλουζάκια, με ντουντούκε. είναι έξω από τα εκλογικά τμήματα και κάνουν την προεκλογική του εκστρατεία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι όμω θέμα ενό κόμματο. όλοι το κάνουν απολύτω. Ε, και κάτι άλλο που είπαμε κι εμεί υπήρχαν πολίτε οι οποίοι, ε, ε, έτσι, όχι, όχι κομματικοποιημένοι, χωρίς κανένα πολιτικό έτσι, χρωματισμό ή ε, προτιμήσεις. Αλλά πολλοί πολίτες έδιναν εξουσιοδότηση και δεν, μάλλον, και δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Γιατί? Υπάρχει Μάλλον δεν ήταν, όχι, δεν ήταν ξουδότηση, ήταν ε, οι πολίτε. Υπάρχουν κάποιοι πολίτε που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ω παρατηρητέ στα εκλογικά τμήματα, ε, αλλά πηγαίνουν πρώτα εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, ε, μετά διάφοροι άλλοι αντιπρόσωποι και δεν έχει χώρο για του απλού πολίτε που έχουν δικαίωμα και που του έχουν καλέσει να παρευρίσκονται. Αυτά ήταν τα προβλήματα. Ε, τα αποτελέσματα. Το κόμμα, το δεξί κόμμα, ένα Ε, είδε να αλλάζει η κατάσταση. Μέχρι τώρα στις εκλογές ε, της ε, βουλευτικές κυβερνούσε το μέτωπο. Αυτά. Δεν έχω να σας πω περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις ή άλλα σχόλια. Θα μπορούμε στη συνέχεια να το συζητήσουμε για να τα αναλύσουμε. Τελειώνω, όπως είπα και στην αρχή, με ευχαριστίες για την υποστήριξη. Από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τους παρατηρητές και τα λοιπά. Με μεγάλο επαγγελματισμό και πολύ μεγάλη ευσυνειδησία συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι διαπιστώνω και μου κάνει εντύπωση. Πώς να το πω. Το υψηλό επίπεδο ε, κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας ζητάνε όλοι να πηγαίνουμε για παρατήρηση εκλογών γιατί υπάρχει ένα background, ε, μεγάλη εμπειρία σε πολλές χώρες στη Μοζαμβίκη, ας πούμε, αυτό το καιρό έχουμε παρατήρηση εκλογών, αλλά σε όλο τον κόσμο ζητούν παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε φορά που πηγαίνουμε, και οι κυβερνήσει, τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα επικοινωνία, όλοι γνωρίζουν και σέβονται πάρα πολύ το ρόλο και τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και μα ευχαριστούν. Είναι και ευγνώμονε και μα ζητούν να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή παρατήρηση εκλογών και σε επόμενε εκλογέ. Αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας γιατί είναι επιτυχία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών όργανων. Ευχαριστώ στα ελληνικά, λέει ο εμιλητής πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο. Κύριοι συνάδελφοι, να σα ενημερώσω ότι ο κύριο Λόπε, επικεφαλής τη αποστολή, δεν μπορούσε να είναι σήμερα στην Επιτροπή μα αλλά θεωρώ ότι ο κύριος συνάδελφος έκανε μια πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών στη... στο Ελσαλβαδόρ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην αυτοεξοχότητα, στην πρέσβη της, ε, του Ελσαλβαδόρ, στην κυρία Βιλατόρο, να μας πει εκείνη τα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχετε και χαιρετισμούς ε, και ε, προς όλους τους βουλευτές, ε, τον κύριο Ιτουργάης και όλα τα μέλη και σε υπηρεσίε εξωτερική δράση, εξοχότατοι, διπλωματικοί εκπρόσωποι, πρέσβει, αξιότιμε κυρίε και κύριοι. Καταρχά, θα ήθελα βέβαια να σα ευχαριστήσω για αυτά που είπατε και κυρίως την πρόσκληση που μου στείλατε για να παρευρεθώ. Ευχαριστώ την πρόεδρο Σακοράφα. Ε, είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνεδρίαση επανειλημμένα για διάφορους λόγους χρονικούς, προγράμματος, δεν καταφέραμε να βρεθούμε και τελικά σήμερα συνεδριάζουμε για το σκοπό αυτό. Όπως είπε ε, ο κύριος Ιτουργκάης και τον ευχαριστώ πολύ για την ε, πλήρη του έκθεση για τις εκλογές που έλαβαν χώρα στο Σαλβαδόρ στις 4 Μαρτίου. και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές πρέπει να πούμε, και το λέω αυτό με μεγάλη ικανοποίηση, ότι οι εκλογές αυτές ε, που ήταν και ε, δημοτικές και βουλευτικές έγιναν με μεγάλη ειρήνη, με ελευθερία της έκφρασης και σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Το Ελσαλβαδόρ είναι μια νέα δημοκρατία, νεαρή, και έχουμε ε, προτεραιότητα την εδραίωση των θεσμών, τη διαφάνεια και το σεβασμό των ε, εκλογικών ε, νόμων με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η χώρα πραγματικά αγκάλιασε τους διεθνείς παρατηρητές που ήρθαν στις 4 Μαρτίου για την παρατήρηση των εκλογών. Ήταν πάνω από 2.000 οι παρατηρητές αυτών των εκλογών. 1.700 εθνική και 900 διεθνής. Αυτό σίγουρα επέτρεψε την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών με μεγαλύτερη διαφάνεια, νομιμοποίηση και αξιοπιστία. Υπό την έννοια αυτή, δράτω με τις ευκαιρίες για άλλη μια φορά για να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όλα τα θεσμικά οργανά, το Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους λοιπούς φορείς για τη συμμετοχή τους στις εκλογές αυτές. Με την παρατήρηση των εκλογών, αλλά και όλη την προεργασία που έγινε, έτσι ώστε να γίνει σοβαρή δουλειά και στις 14 διαπερίσματα της χώρας, στις διάφορες επαρχίες. Μέχρι και στο τελευταίο χωριό ε, είχαμε διεθνή παρουσία και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Επιπλέον πρέπει να πω ότι η δουλειά της αποστολής αυτής χαρακτηρίστηκε όχι απλώς από την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα στην παρατήρηση των εκλογών, αλλά και από την αποτελεσματικότητα ε, και τη διαφάνεια. Είμαστε βαθιά πεπισμένοι ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη πραγματογνωμοσύνη στην παρατήρηση των εκλογών. Χαιρόμαστε για την τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Ο κύριος Ιτουργάης αναφέρθηκε ε, σε συντομία στα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν την ημέρα των εκλογών. Και θα ήθελα να πω και εξ ονόματος της κυβέρνησης του Ελσαλβαδόρ ε, θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυτές τις συστάσεις και τα συμπεράσματα έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επόμενες εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι οι συστάσεις αυτές θα μας επιτρέψουν ε, να εδραιώσουμε το εκλογικό σύστημα, να βελτιώσουμε το πολίτευμα για να ε, αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η δημοκρατία στη χώρα μας. Η κυβέρνηση του Ελσαλβαδόρ ελπίζει να μπορεί να υπολογίζει στη συνεργασία και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, βελτιωθούν τα μέτρα που θα πάρουν. Και πριν ε, τελειώσω θα ήθελα να επαναλάβω ότι το El είναι στη διάθεσή σας ε, να υποδεχτεί ε, αποστολές παρατήρησης εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Στις 3 του Φλεβάρι το 2019 θα διεξαχθούν προεδρικές εκλογές και ελπίζουμε να έχει συμμετοχή και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή για να κάνουμε την προεργασία και την προετοιμασία, την επιμελητία για να έρθει η αποστολή. Περιμένουμε λοιπόν να έχουμε αντίστοιχη συμμετοχή στο άμεσο μέλλον. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή σχόλια που μπορεί να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πρέσβη και θα δώσω τώρα το λόγο στην προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στη Διεύθυνση για την Κεντρική Αμερική, στην κυρία Αφέλτ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Επειδή μετά από την υπηρεσία παρατήρησης, εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ θα γίνουν σχόλια από τη συνάδελφο την ίδια για την αποστολή, εγώ να μιλήσω για το γενικό πλαίσιο, την κατάσταση όπως βλέπουμε να δημορφώνεται στο μέλλον. Θέλω επίσης να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου για όλους όσους μετήχαν και έκαναν την αποστολή αυτή μια επιτυχημένη αποστολή. Τον ε, πρέσβη Βιλατόρο, την πρέσβη Βιλατόρο μάλλον, τον πρέσβη, τον επικεφαλής της αποστολής παρατήρησης και όλα τα μέλη της αποστολής αυτής. Σας ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι αυτή η αποστολή εκλογική παρατήρηση είχε μεγάλη σημασία για την ενίσχυση τη αξιοπιστία του εκλογικού συστήματο στη χώρα, άρα και την εμπιστοσύνη στου δημοκρατικού θεσμού. Αυτό για μα είναι βασική σημασία για μια κοινωνία με τόση πόλωση για τόσα πολλά χρόνια. Η εμπιστοσύνη στη λειτουργία του δημοκρατικού συστήματο και τον δημοκρατικό διάλογο επιτρέπει στην κοινωνία να ε, ξεπεράσει τα προβλήματα με την επίτευξη πλειοψηφία. Αυτό ε, θα ισχύει και για το Σαλβαδόρ. Ε, επίσης, για τον εθνικό διάλογο τα τελευταία χρόνια για την ασφάλεια των πολιτών, την παιδεία, το περιβάλλον και το κατά πόσο είναι ευάλωτη όλη η κοινωνία είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να πετύχουμε εθνική συνένεση σε τέτοιες περιπτώσεις γύρω από την κεντρική κυβέρνηση. Καλωσορίζουμε την συμφωνία του φετινού Ιουλίου που επετέχθη μεταξύ των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στην ε, Βουλή για συνένεση σε πέντε τομείς προτεραιότητα, δηλαδή ασφάλεια, δημοκρατικούς θεσμούς, ανάπτυξη, εκπαίδευση και υγεία. Η προθυμία να βρεθούν σε μια σύγκληση μεταξύ των πολιτικών ε, φορέων και συμμετεχόντων στην πολιτικό βίο είναι ε, καθοριστικά για να δούμε αν θα πετύχουν οι πολιτικές διαδικασίες και οι μεταρρυθμίσεις και το κατά πόσο θα μπορέσει όντως η κοινωνία να ξεφύγει από την πόλωση που προανέφερα. Το Σαλβαδόρ πέτυχε πρόοδο από το τερματισμό των εμφυλίων συγκρούσεων και την πολιτική συμφιλίωση. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί εύρωστοι δημοκρατική θεσμή που παίζουν ζωτικό ρόλο στην εδραίωση αυτής της διαδικασίας. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρές δυσκολίες για τη χώρα ως προς την συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη και την ασφάλεια των πολιτών. Εμείς, ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουμε τη χώρα στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι λόγου χάρη η υποστήριξη προς το πλάν σεγκούρο στο Σαλβαδόρ. Δηλαδή το πρόγραμμα για την ασφάλεια στο Σαλβαδόρ. Ε, είναι δύσκολη καιρή, αλλά παρά τα εμπόδια μπορέσαμε χάρη στη συνεργασία μας να οργανώσουμε και μια καλή συνεδρίαση του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη ΣΕΛΑΚ και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Και εμεί σα ευχαριστούμε και θα δώσω το λόγο στην ε, προϊσταμένη τώρα στην υπεύθυνη του τμήματο εκλογική παρατήρηση τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, την κυρία Ντελαπουέντε. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ιτουργάης ήδη ε, αναφέρθηκε στη σημασία ε, των αποστολών εκλογικής παρατήρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο, πόσο ε, καλά καταρτισμένες είναι και ε, επαγγελματικές. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα ήθελε με τη σειρά της να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη στις αποστολές αυτές και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν για την αφοσίωσή τους και το έργο τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Προφανώ και στα πλαίσια τη σημερινή συνεδρία θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Τουργκάιφ και ε, από πλευράς υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, γιατί είναι εξαιρετική η ε, αποστολή και πραγματικά με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή. Γνωρίζετε ότι αυτές οι αποστολές είναι πολύ σημαντικές για διάφορους λόγους. δίνουν μεγάλη ε, ασφάλεια και στον πληθυσμό από την ίδια τους την παρουσία και ε, ε, εξασφαλίζουν και την εκλογική διαδικασία. Και έτσι ηρεμούν και τα πνεύματα κάπως. Όπως γνωρίζετε, σε όλες τις εκλογές μπορεί να υπάρχουν κρίσεις και προβλήματα και εντάσεις ε, και αυτό λοιπόν οι δικές μας ε, αποστολές παρατηρήσεις βοηθούν στο να πέσουν οι τόνοι, να ε, ηρεμήσουν τα πνεύματα. Και, να... στηρίξουμε το σύστημα ώστε να συνεχίσει η ειρηνευτική διαδικασία και η διαδικασία εξέβρεσης πολιτικής συνένεσης. Μια άλλη σοβαρή συνεισφορά της αποστολής εκλογικής παρατήρησης ήταν να προσφέρει επικοδομητική συνεισφορά παρακολουθώντας πώς διεξήχθησαν οι εκλογές, πώς διαμορφώθηκε το όλο σύστημα, πώς διοργανώθηκαν οι υπεύθυνοι με την ε, κατάλληλη προοπτική, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη παρατήρηση και τα απαραίτητα στοιχεία για το πώς έγινε η διεξαγωγή. Ήταν λοιπόν ένα πολύ καλό εργαλείο για τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας στο μέλλον η αποστολή αυτή. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει διαρκής πρόοδος από τη μία από τον ένα γύρο εκλογών στον άλλο. Υπάρχουν 23 συστάσεις, συντάχθησαν μετά την διεξαγωγή των εκλογών, ε, καλύπτουν όλες τις πτυχές της εκλογικής διαδικασίας και να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για το κύριο Τουργκάης ε, κάποια τα ανέφερε, κάποιε από τις αδυναμίες. Οι συστάσεις αφορούν τον, ε, το πώς ορίζονται οι, παρα, για τις παραβιάσει από την πλευρά κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία, το τι γίνεται με την αφορευτική επιτροπή, με την καταμέτρηση των ψήφων, με την περίοδο σιωπή πριν τι ε, ε, εκλογές τη ίδια, όπου εκεί υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, ενίσχυση του σχηματισμού ομάδων, της σύνθεσης μιας εθνικής ομάδας για να συμμετέχουν στην διοργάνωση των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχει βάλει μια νέα φάση σε αυτές τις αποστολές που είναι μια παρακολούθηση πολύ πιο στενή και πολύ πιο βαθιά των συστάσεων και των συμπερασμάτων στην τελική φάση. Ε, έχουμε αυτό που ονομάζουμε τελική επίσκεψη, όπου επιστρέφουμε για να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και να αρχίσουμε να συζητούμε την εφαρμογή τους με τους ενδιαφερόμενους στο Σαλβαδόρ, ενδεχομένως τώρα τις ε, εθνικές αρχές και άλλες αρχές. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιες συστάσεις είναι πιο εύκολες στην εφαρμογή τους και κάποιες άλλες πιο δύσκολες. Οι συστάσεις που συμβαίνουν νομοθετικές αλλαγές βεβαίως είναι πιο βαριές και πιο χρονοβόρες Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε στην υπόθεση, την περίπτωση του Σαλβαδόρ, είναι ότι στο παρελθόν και σε άλλες αποστολές που είχαμε, είδαμε ε, ένα ενδιαφέρον από πλευράς των αρχών της χώρας να εφαρμόσουν τις συστάσεις και τις ε, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2018 ε, μετά τις εκλογές, στο τέλος των εκλογών συνταθήκαμε και με εθνικούς φορείς και με διεθνείς συντάχθηκε ένας οδικός χάρτης για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πρέσβη για τα λόγια της, ότι θα ασχοληθούν με την υλοποίηση. Η δική μας αντιπροσωπεία επίσης εκεί βοηθάει, συνεργάζεται με τους διαφόρους αρμοδίους φορείς έτσι ώστε να δώσουμε μια συνέχεια και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε πιο πρακτικό και αν χρειάζονται κάποια τεχνική βοήθεια, αν υπάρχει κανένα αίτημα για συνδρομή ε, Πολύ ευχαρίστω. Αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι όπως και στο παρελθόν το Σαλβαδόρ θα μελετήσει αυτές τις συστάσεις και θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του το 2018 και μπορούμε εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Σακορά. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους μας τους προσκεκλημένους και την πρέσβυρα του Σαλβαντόρ, τον κύριο Ιτουργκάης και την εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ και την τελευταία εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ που μας ε, μίλησε για την τόσο ακριβή επισκόπηση που έγινε για την εκλογική διαδικασία. Και ήθελα και να ευχαριστήσω, να εκφράσω και τι ευχαριστίε μου και τη χαρά μου που ακόμη και δεν είχα την διερμηνία από τα Ιταλικά στο πρώτο κομμάτι της συνεδρίασης. Ε, χαίρομαι που τώρα ε, έχω καταφέρει παρόλα αυτά να καταλάβω τη θετική ε, κατάσταση σε σχέση με τις εκλογές και υποδοχή των ε, διεθνών παρατηρητών ήταν ε, θετική και μεγάλη προσπάθεια έγινε για να, τηρηθεί, να τηρηθούν οι κανόνες, να υπάρξει διαφάνεια και ε, ανεξάρτητη και δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών από την πλευρά τη κυβέρνηση, των θεσμών και το καθεξή. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν παρατυπίε ή παρανομίε σοβαρέ, σοβαρά προβλήματα ή τριγμοί. Ωστόσο, ένα από τα πράγματα που με εξέπληξαν είναι ότι οι δυσκολίες υπήρξαν από το δικαστήριο ε, για να ελέγξει το κατά πόσο ήταν νόμιμες οι χρηματοδοτήσεις. Δεν το κατάλαβα πολύ καλά γιατί δεν υπάρχει εδώ νόμος. Και ήθελα να θέσω μια ερώτηση κάπως γενικότερη. Οι εκλογέ αυτές που διεξήχθησαν σε ένα κλίμα γενικώ θετικό θα έλεγα. Και αν δεν κατάλαβα άσχημα, με σημαντική συμμετοχή των πολιτών έγιναν σε κλίμα σεβασμού των συστάσεων που έχουν εκδώσει οι διεθνείς οργανισμοί. Οπότε, η παρατήρησή μου είναι γενικότερη. Ας ελπίσουμε ότι πρόκειται ε, για την έναρξη μιας ε, διαδικασίας αλλαγής της πολιτικής νοοτροπίας στη χώρα, σεβασμού των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, ε, συμφιλίωσης και συνένεσης. Μπορεί να είναι πραγματικά η αρχή μιας νέας πορείας σε σχέση με τα δικαιώματα σε μια χώρα που κάνει τεράστιε προσπάθειες, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, για να επιταχύνει την πρόοδο προς τον σεβασμό των ελευθεριών και των δικαιωμάτων. Ίσως λοιπόν στι επόμενε εκλογέ, όπως υπενήχθηκε η πρέσβυρα, θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω τεστ και έλεγχο του κατά πόσον αυτή η διαδικασία αλλαγή ε, πορεία τη χώρα προχωρεί. Αυτή ήταν η γενική μου παρατήρηση να προσπαθήσουμε λίγο να προβάλλουμε τις θετικές εξελίξεις στο μέλλον, υπό το φως των πορισμάτων, που θεωρώ ότι είναι ευχάριστα ε, από την όλη προσπάθεια παρατήρησης των εκλογών. Και πάλι λοιπόν ευχαριστώ για τις τόσο λεπτομερείς πληροφορίες που μας δώσατε, ήταν κατατοπιστικότατες και μπράβο σε όλους για την αφοσίωσή τους, αυτούς που πήγαν ως εκεί και παρατήρησαν με τόσο μεγάλη επιμέλεια την διεξαγωγή των εκλογών. Ευχαριστώ. Κύριος Μάτο, Αντιπρόεδρος, έχει το Ευχαριστώ Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την πρέσβη ε, και σένα Κάρλος και την Κόντσα. Ακούσαμε τις παρατηρήσεις, τις εξηγήσει, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ε, πρέπει να σας πω ότι εμένα μου αρέσει πολύ να ακούω τέτοια λόγια για χώρες της Κεντρικής Αμερικής ε, όπως το Σαλβαδόρ που κάνει μεγάλες πρόοδους. Βέβαια πάντα χωράει βελτίωση και κάτι έχει επομείνει για να βελτιωθεί ε, ε, όλοι θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Το, αυτό το ασφαλές Σαλβαδόρ ε, είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε διακάως. Και σίγουρα οι συστάσεις θα υλοποιηθούν, είμαι βέβαιος, και θα λειτουργήσουν. Και κάτι που με χαροποιεί ακόμα περισσότερο εμένα είναι ότι συνεχίζουν να ποντάρουν και να πιστεύουν ε, στις αποστολές εκλογικής παρατήρησης. Όταν είναι σωστές οι εκλογές, ε, δίκαιες, ανώθευτες, γίνεται σεβαστός ο νόμος και το Σύνταγμα. Δεν φοβάται κανείς να προσκαλέσει εκλογικούς παρατηρητές για να βοηθήσουν και να συνεργαστούν με ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μου άρεσε πολύ η σημερινή συζήτηση αυτά που άκουσα και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν είναι πάντα εύκολη η μετάβαση, όπως είπαμε, στα θέματα της ασφάλειας, αλλά ε, σίγουρα έχετε πάντα στο πλευρό σας ε, το Κοινοβούλιο και την αντιπροσωπεία μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε συνάδελφοι. Θέλετε, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, ναι, Ευχαριστώ. Εσύ ναι. Δύο σχολεία με την άδεια της Πρόεδρου μας και απαντώντας στην κυρία Κινίτσι για τη χρηματοδότηση. Είναι γεγονός ότι στο θέμα της χρηματοδότησης υπήρχαν δύο σημεία που θα ήθελα να σας εξηγήσω με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι στην εισαγωγή μου. Το εκλογοδικείο, Electoral, ε, εξέφρασε καταγγελίες και παράπονα. Θέλανε να δούνε χρήματα από τον προϋπολογισμό, τον κρατικό. Είχαν ζητήσει ε, χρηματοδότηση αλλά η Βουλή δεν την ενέκρινε. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν 100% με τον τρόπο που θα ήθελαν. Ήθελαν μια χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των εκλογών και δεν τα κατάφεραν ε, για να διεξαχθούν πιο απρόσκοπτα οι εκλογές και να είναι η δουλειά τους ακόμα καλύτερη. Και παρά το γεγονός όμως δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για το δικαστήριο αυτό, ότι τα κάνανε πολύ καλά. Τα βγάλανε πέρα με τα λιγότερα λεφτά που τους ενέκριναν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα για την άλλη φορά, γιατί θα του πούνε ότι ορίστε με αυτά που σας δώσαμε τα βγάλατε θαυμάσια πέρα γιατί θέλετε περισσότερα. Ε, ήταν πραγματικά υποδειγματικές αυτές οι εκλογές για όλη την ε, περιοχή και για όλους εμάς. Ακούσαμε ότι η χώρα αυτή είναι νεαρή νέο σύστατη έχει γνωρίσει τραγωδίες τρομακτικές και συμφορές και δεινά και αυτή η μετάβαση ε, σε αναζήτηση της ειρήνης και στο δρόμο προς τη δημοκρατία είναι κάτι θαυμάσιο. Και ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές και θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε εκείνους που δίνουν το παράδειγμα και στη Λατινική Αμερική και στον κόσμο ολόκληρο, φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές ε, και, και χωράνε βελτιώσεις. Δεν είπε κάνει ότι είμαστε τέλειοι. Αλλά πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο η χώρα. Το δεύτερο. Σε σχέση με τις προηγούμενες ευχαριστίες, είπε και ο συνάδελφος Μάτο για το πόσο σημαντικέ είναι αποστολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι άλλο που ξέχασα, οι πρέσβεις μα εκεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ανδρού Γκασόλ, για να το πω με το όνομά του, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, υποστήριξη, επιμελητεία, βοήθεια γενικότερα και τους άλλους πρέσβεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας. Αυτοί οι πέντε είναι. Έχουμε εκεί πρεσβείες και έκτος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουν ανεξαιρετική δουλειά. Μας εξήγησαν τι είναι η χώρα, τι συμβαίνει, με εξαιρετικές ενημερώσεις, ε, τι περίμεναν ε, κλπ. Ευχαριστώ. Gracias. Ε, ευχαριστώ με την άδειά σα, ε, Πρόεδρε. Σύντομα, δεν θέλω παρά να σας ευχαριστήσω και πάλι για τα καλά σας λόγια, για τα σχόλιά σας. Και όπως είπατε, κύριε Μάτο, βεβαίως υπάρχουν πράγματα που χωράνε βελτίωση. Είναι μια διαδικασία αυτή και η διαδικασία γίνεται βήμα-βήμα. Το σημαντικό είναι να έχεις το όραμα, να θέλεις να βοηθήσεις, να βελτιώσεις και να συνεχίσεις σε αυτή τη δημοκρατική ε, οδό, όπως είπε και ο κύριος Σιτουργκάης. 26 χρόνια έχουν περάσει από τότε που υπογράψαμε τις ειρηνευτικές συμφωνίες μόνο και θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε ως έθνος και ως χώρα σε αυτή την κατεύθυνση. Και συμφωνώ με τον κύριο Τουργάης. Ο δικός σας πρέσβης εκεί ο Αντρούμπα Σόλς ε, είναι πολύ ε, αξιόλογος και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και η πρεσβεία μου και η κυβέρνηση. Σύμφωνο και με εσάς κύριε Μάτο και με τους υπαλλήλους υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε στην εκλογική διαδικασία, στην παρατήρηση των εκλογών και αυτό είναι επιθυμία του λαού ολόκληρου να προχωρήσουμε στη δημοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η αποτίμηση λοιπόν των εκλογών, κύριοι συνάδελφοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι απόλυτα θετική. Αναφέρθηκε πάρα πολλέ φορέ η λέξη υπόδειγμα και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε αυτό από τον συνάδελφο, ο οποίο ε, ε, πήγε σαν παρατηρητή ε, στη συγκεκριμένη χώρα. Ε, και εμεί, σαν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε το λαό της, του Ελ Σαλβαδόρ για την υπεύθυνη και δημοκρατική στάση που κράτησε σε όλη την διαδικασία των, των εκλογών. Τώρα τα προβλήματα που έχουν ε, επισημανθεί νομίζω ότι είναι στη διαδικασία του να βελτιωθούν, ούτω ώστε να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του, του λαού του Ελ Σαλβαδόρ στην εκλογική διαδικασία αλλά και στου θεσμού. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο συνάδελφο για την ενημέρωση που μα έκανε, την κυρία Πρέσβη και τις εκπροσώπους τη επιτροπή εξωτερική δράση. Τώρα, παρακαλώ. Να πάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική κατάσταση στην Ικαράγουα. Κυρία συνάδελφε, ξέρω ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγετε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Okay. <laughs> I know, I know οι συνάδελφοι κατά την τελευταία συνεδρίαση τη αντιπροσωπεία τη 5 Ιουλίου δεσμεύτηκαν να, να πραγματοποιηθεί μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Νικαράγουα. Η Νικαράγουα έχει από τον Απρίλιο του 2018 βιώσει σοβαρέ αναταραχέ και μεγάλη κλίμακα διαμαρτυρία. Μέχρι το τέλο του Αυγούστου, 325 άνθρωποι περίπου έχασαν τη ζωή του σε συγκρούσει μεταξύ διαδηλωτών, δυνάμεων ασφαλεία και παραστρατιωτικών ομάδων. Ορισμένε οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν μιλήσει ακόμη και για θάνατο περίπου 450 ανθρώπων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 22 αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω ταραχών. Όπω ήδη γνωρίζετε, οι αναταραχέ αυτέ ξεκίνησαν στι 18 Απριλίου του 2018 σαν διαμαρτυρία ενάντια στη μεταρρύθμιση του συστήματο κοινωνική ασφάλιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αν και ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα απέσυρε την αμφισβητούμενη αυτή μεταρρύθμιση στις 2 Απριλίου, 22 Απριλίου, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν. Τους μήνες που ακολούθησαν, οι διαδηλώσεις οξύνθηκαν και έλαβαν πιο βίαιο χαρακτήρα, θέτοντα το επίκεντρο των ετοιμάτων του στην παρέτηση του Προέδρου Ορτέγκα και την ενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είχε εγκατασταθεί στην Ικαράγουα κατόπιν πρόσκληση τη κυβέρνηση, κλήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Η απόφαση τη κυβέρνηση Νικαράγουα να τερματίσει την παρουσία τη αποστολή του ΥΠΑ του Αρμοστή στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αντίθετη με το στόχο τη πλήρου λογοδοσία για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη παροχή δικαιοσύνη στα θύματα τη βία. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα τη έκθεση αποστολή του ΥΠΑ του Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να επαναξεταστούν από τι αρμόδιε αρχέ τη χώρα και να ληφθούν μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων τη έκθεση να σας υπενθυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή και σαν πρόεδρος του ΔΕΚΑΜ καταδίκασα τη βία που είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπινων ζώων. Η βία δεν αποτελεί λύση και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο ανοιχτό και χωρί περιορισμού διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί τη μόνη λύση. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν πλήρως και να παρέχουν πρόσβαση στις αποστολές της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα μου επιτρέψετε τώρα να δώσω το λόγο στην αυτοεξοχότητα των τη της Νακαράγουα, τον κύριο Σαντίνο Μόντες, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Σοφία Σαχοράφα, πρόεδρε της ΔΕΚΑΜ, αξιότιμα μέλη της αντιπροσωπείας, αξιότιμοι βουλευτές, συνάδελφοι πρέσβεις της Κεντρικής Αμερικής και διπλωματικοί υπάλληλοι, αξιότιμοι και αγαπητοί φίλοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αγωνίζεστε μαζί μας για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία στην Ικαράγουα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον της αντιπροσωπείας σας και ιδιαίτερα της Προέδρου στις εξελίξεις της δημοκρατικής διαδικασίας ε, στη χώρα. Η κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης και Ενότητας υπό την ηγεσία του Προέδρου ε, Κομμαντάντε Ντανιέλ Ορτέγα έχει πάει για επικοινωνία με το Ευρωκοινοβούλιο βασιζόμενη στο σεβασμό πιστεύουμε ότι ο διάλογος βοηθάει στην ε, κατανόηση των λαών μας. Η κυβέρνηση της ε, Νικαράγουας εγγυάται την νομιμότητα και τους δημοκρατικούς μηχανισμούς που έχει επιβάλει το Σύνταγμα και ο νόμος της χώρας, δηλαδή η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας. Από τον Απρίλιο φέτος η Νικαράγουα έχει αναγνωριστεί ότι αναπτύσσεται οικονομικά. Τα τελευταία επτά ετία είχαμε αύξηση 5% του ΑΕΠ. Και αυτό κατέστη δυνατό λόγω και των κοινωνικών προγραμμάτων. Το 2007 η φτώχεια αφορούσε το 47% του πληθυσμού, ενώ σήμερα αυτό έχει μειωθεί στο μισό. Γύρω στο 22% είναι η φτώχεια στη χώρα. Το ίδιο ισχύει και με την ψαλίδα ε, πλουσιωτέρων και φτωχοτέρων. Το έχουμε μειώσει κατά 50% αυτό το χάσμα, τη διαφορά. Ήταν η δεύτερη ασφαλέστερη χώρα σε όλη τη Λατινική Αμερική και σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε σαν νησίδα ε, ασφαλείας στην περιοχή. Η Νικαράγουα είναι έκτη ε, στην Παγκόσμια Κατάταξη Ισότητας Φύλων το 2017. Αυτό το λέει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και είναι στο 10 ε, ήταν στη δέκατη θέση, ενώ σήμερα έχει φτάσει στην έκτη. Είναι από τη Λατινική Αμερική η χώρα με τη μεγαλύτερη ισότητα, μετά την Ισλανδία, Νορβηγία, Φινλανδία, ε, Ολλανδία και Σουηδία έχει κλείσει η ψαλίδα της διαφοράς του φύλου κατά 80% και πλέον. Οπότε, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί τομείς που δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εύνοια των πολιτών ανδρών και γυναικών στην Νικαράγουα και που τις χρηματοδοτούν με ανήθικο τρόπο ξένες δυνάμεις από το 2007 ήρθαν να κάνουν πραξικόπημα. Αυτοί που λέγονται τώρα οι ήπιοι οι μαλακοί για να ρίξουν την κυβέρνηση που έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει εκλεγεί ελεύθερα και δημοκρατικά. Τρει μήνε πραγματικά ζήσαμε ε, ένα πραξικόπημα, μια απόπειρα πραξικοπήματο με βία, με υποδάβληση μίσου, με παραπληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωση, με χειραγώγηση που την προετοίμαζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό με στόχο να δημιουργήσουν μια αρνητική διεθνή κοινή γνώμη απέναντι στην κυβέρνηση του Προέδρου Κομαντάντε Ντανιέλ Ορτέγα για να τον καταδικάσουν και να τον απομονώσουν διεθνώς με συνοδεία κυρώσεων που ε, θα πλήξουν το λαό και μόνο και τις οικογένειες. Ο πρόεδρος, ο ε, κομμαντάντε Ντανιέλ, αποφάσισε να συγκαλέσει εθνικό διάλογο για να ξεπεράσουμε αυτή την πολιτική κατάσταση. Ε, παρόλα αυτά, την πρώτη μέρα του διαλόγου, όταν του ζήτησαν του κομμαντάντε Ορτέγα να μαζέψει την αστυνομία ε, στα στρατόπεδα το έκανε 15 μέρες χωρίς να τους αφήσει να βγουν έξω ας πούμε στη Μασάγια και στο Ινοπέτεπε και στην Εριάμπα όπου καθημερινά υπήρχαν ομάδες τις νύχτες με τηλεβόες για να ε, υβρίζουν τους αστυνομικούς και όχι μόνο αυτό, τους πυροβολούσαν κιόλας ε, με μολότοφ, με όλμους, με πυροβόλα όπλα και υπήρξαν και τραυματίες αστυνομικοί. Δεν ήταν καθόλου φοιτητέ, εγκληματίες, ήταν και σικάριος, πληρωμένοι δολοφόνοι ε, για να δημιουργήσουν αυτά τα οδοφράγματα και να μην αφήνουν το λαό να κυκλοφορεί ε, ε, ελεύθερα. Ο κομμαντάντε Ορτέγα το κράτησε το λόγο του. Υπάρχει ο σύντροφος Φρανσίσκο Αράους, που είναι γιος δύο ιστορικών στελεχών των Σαντινίστας, αγωνιστών, και ήταν θύμα. Ο πατέρας του επίσης είχε δολοφονηθεί από την πολιτοφυλακή του Σομόσα. Ενώ η μητέρα του που ζει ακόμα είναι η ροήδα της Νικαράγουας, όλη της τη ζωή έχει αγωνιστεί και ε, είναι γνωστή ως η αγρότησα του Κουά, που είναι μια επαρχία στο βορρά της χώρας. Μετά από τέτοια βία, ένα σημαντικό τμήμα του λαού είχε τρομοκρατηθεί και υπήρξε ε, τρομοκρατική ε, εκστρατεία, τρομοκράτηση του λαού από το διαδίκτυο, από τις τηλεοράσεις, όπου έδειχναν όλες αυτές τις βαρβαρότητες που έκαναν στους αντινίστας αυτή η τύπη. Με στόχο ε, να τρομάξουν το λαό. Και ο λαός δεν ήξερε τι να κάνει. Τέλος, αναγκάστηκαν να μείνουν τρεις ε, μήνες στα σπίτια τους κλεισμένοι χωρίς να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και ο κόσμος άρχισε μετά σιγά σιγά να βγαίνει. Οι σαντινίστας και οι πολίτες ε, ε, χρησιμοποιούν το δικαίωμα που τους επιτρέπει να βγουν στο δρόμο και να ανακτήσουν τη φυσιολογική ζωή στη χώρα. Άρχισε ο λαός να απαιτεί να βγει αστυνομία στο δρόμο και άρχισαν από κοινού λαός και αστυνομία να ε, διαλύουν τα οδοφράγματα και τελείωσε αυτή η υπόθεση. Στην Ικαράγουα υπάρχει μια διαδικασία ε, δημοκρατική που γίνεται σεβαστή. Ναι στη συμφιλίωση, όχι στην ατιμορρησία. Δεν είναι το, το ίδιο πράγμα. Οι εγκληματίες που έχουν κάνει δολοφονίες θα πρέπει να υποβληθούν ε, και στον νόμο και να υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι από τον Οκτώβριο του 2016 συζητούμε ε, με τους αρμόδιους ε, φορείς για να αναθεωρήσουμε τον εκλογικό μας νόμο. Δεν τα έχει ορίσει η κυβέρνηση αυτά, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο. Υπάρχουν πράγματα που χωρούν βελτίωση, βεβαίως και το κάνουμε και με την ε, ε, οργάνωση ε, ΟΕΑ την Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών και καλούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας βοηθήσουν για τον εκδημοκρατισμό της χώρας μας. Για την ειρήνη και την ασφάλεια που τόσο επιθυμούμε και που θέλησαν να μας καταστρέψουν. Ευχαριστώ πολύ. Και σα ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη και θα δώσω το λόγο στην υπηρεσία εξωτερική δράση, την κυρία Άφελτ. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ πολύ. Ίσως κινδυνεύω να επαναλάβω κάποια από αυτά που ήδη υπόθηκαν. Η δική μας αντίληψη της όλης κατάστασης στην Ικαράγουα έχουν περάσει πέντε μήνες από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση. Η κατάσταση ανησυχεί πολύ. Δεν είναι κρυφό αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάνω από 322 500 θύματα ε, σε στιγμές που γίνονται διαδηλώσεις ή και άλλες στιγμές στράφηκαν δημόσιες αρχές κατά των ε, διαδηλωτών, αλλά κυρίως είναι αρχές διοκτικές, αυτές που έχουν προκαλέσει τους θανάτους και άλλες οργανωμένες ομάδες. Υπάρχουν αρκετοί που βρίσκονται σε κράτηση. Οι αριθμοί τη κυβέρνηση λένε ότι είναι 204 άτομα, αλλά ο ειδικό μηχανισμό παρακολούθηση για την Νικαράγουα λέει ότι είναι 320 οι κρατήσει τουλάχιστον. Η κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ένα κύμα ποινικών διώξεων κατά των ομάδων της αντιπολίτευσης με την εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου ως πρόσχημα και αναφέρονται πολλές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έλλειψης νόμιμης εκδίκασης των υποθέσεων. Η κρίση στην Ικαράγουα Επίσης, έχει απτές συνέπειες στην οικονομία και την, ε, τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Ακούμε εκτιμήσεις ότι είναι 30.000 οι πολίτες της Νικαράγουας που εγκατέλειψαν τη χώρα. Πηγαίνουν κυρίως προς την Κωνσταντίνα. είναι περίπου 300.000 έως 500.000 αυτοί που έχασαν τη δουλειά τους και τον Ιούνιο είχε κάμψει 12% η οικονομία. Η ανάπτυξη που ήταν συνήθως 5% προβλέπεται στο μείον 4% σε σχέση με τη μέση ανάπτυξη ε, που γνωρίζαμε. Επίσης τα κεφάλαια ε, φεύγουν από τη χώρα και οι ξένες επενδύσεις έχουν κατρακωθεί με το ξέσπασμα της κρίσης. Το εμπόριο, υπηρεσίες και ο τουρισμός λοιπόν έχουν πληγεί δραστικά. Όλοι οι τομείς έχουν πληγεί ιδιαίτερα, ενώ κάποιοι τομείς που εξαρτώνταν από τις εξαγωγές και στρέφονταν κυρίως προς τις εξαγωγές, κάπως έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν. Επίσης, ακούμε, το ανέφερε και ο πρέσβης, ότι ανέφερε ότι το περιβάλλον είναι σχετικά ασφαλή στη χώρα. Εμείς ακούμε ότι η εγκληματικότητα διωγγώνεται. Υπάρχει σοβαρή πόλωση στη χώρα. Ο πρόεδρος καταδίκασε τις εκκλήσεις και απέρριψε τις εκκλήσεις για πρόορες εκλογές ή για την έναρξη εθνικού διαλόγου. Η αντιπολίτευση ζήτησε πανεθνική πανικαραγουανή ανεργία, ε, για χθε, Πράγμα που ε, δεν έχει γίνει από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Η κατάσταση λοιπόν αλλάζει μέρα με τη μέρα και έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας με τουλάχιστον 8 δηλώσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε επίσης εκφράσει τις ε, ανησυχίες μας διμερώς με, σε εκπροσώπους της κυβέρνησης και άλλους ενδιαφερομένους και έχουμε καταστήσει σαφές ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πραγματικά απευθύνουμε στεναρή έκκληση προς την, για την έναρξη διαλόγου εθνικής συμφιλίωσης. Πριν το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεκλήθη από την κυβέρνηση να στηρίξει ακριβώ μέρος αυτού του εθνικού διαλόγου και, ο, και είπατε εκπρόσωπο. είπατε εκπρόσωπο και απαντήσει στον Υπουργό Εξωτερικών τη Νικαράγουα ότι θα στηρίξει την διαδικασία και οικονομικώ. Ένα πακέτο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν προβλεφθεί για να υποστηρίξουμε τις δύο επιτροπές που είχε οργανώσει η Διαμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την Ικαράγουα συγκεκριμένα με την ε, παρακολούθηση του κυρίου Μεσένη και με την ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων να παρακολουθούν την εκταμείευση των ποσών. Επίση, τα κονδύλια αυτά ήθελαν να στηρίξουν το ρόλο διαμεσολάβηση τη Καθολική Εκκλησία, που υποτίθεται ότι θα αναλαμβανόταν από την Καθολική Εκκλησία στην διαδικασία του διαλόγου. Και έχουμε οργανώσει και το σχετικό χαρτοφυλάκιο με το πώ θα ενημεθούν τα ποσά για να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται πραγματικά οι πολίτε τη χώρα. Με άλλου διεθνεί και περιφερειακού εταίρου συνεχίζουμε να πιέζουμε, να ασκούμε πιέσει για την έναξη διαλόγου εθνική συμφιλίωση, γιατί πιστεύουμε ότι είναι η μονή διέξοδο από την κρίση. Βλέπουμε και θα δούμε τι ερχόμενε εβδομάδε αν μπορεί αυτό να γίνει. σω με κάποιο σχηματισμό κάποια μορφή που θα επιτρέψει να ξεκινήσει κάποιο είδου οικοδόμηση συνένεση στη χώρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ και εμεί. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε συνάδελφε, κάποια τοποθέτηση. Ναι, ο κύριος Μάτο, ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Πρέσβη και την ε, Υπηρεσία εξωτερική Δράσης. Κύριε Πρέσβη, πρέπει να αναγνωρίσω ότι όταν ε, αρχίσατε να μιλάτε, ε, πίστευα ότι κάνετε προσπάθειες να βελτιώσετε τη δημοκρατία στην Ικαράγουα και αυτό πραγματικά με ενέπνευσε και, και μου άρεσε, αλλά απογοητεύτηκα γρήγορα ε, στη συνέχεια. Ε, εξαφανίστηκε αυτό το ευχάριστο συνέστημα, γιατί φαίνεται ότι μιλάμε για διαφορετική πραγματικότητα, αυτή που μας περιγράφεται και αυτή που έζησα εγώ, που μελέτησα και που διάβασα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Νικαράγουα ζει σε ανώμαλες περιστάσεις εδώ και καιρό. Το 2007 ε, έγιναν τρεις εκλογές για να εκλεγεί ο πρόεδρος, ενώ ε, Τρει θητείε. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορεί να επανεκλεγεί. Παραβιάστηκε το εκλογικό σύστημα. Και αυτό έτσι κι αλλιώ ε, αυτό είναι σοβαρό, αλλά πιο σοβαρά είναι τα στοιχεία, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε μετά ποιο στέει, να το βρούμε εύκολο είναι να αποδίδει ευθύνε και να μην ε, κοιτάς τι γίνεται στη χώρα. 350 διδολοφονημένοι, πάνω από 2.000 τραυματίες, 700 σε αυθαίρετη σύλληψη. Η ελευθερία της έκφρασης προφανώς απέχει πόρο από το να υπάρχει στη χώρα. Ένας δημοσιογράφος, ο Άγχελ ε, δολοφονήθηκε όταν ε, παρουσίαζε τις ειδήσει ένα πρόγραμμα. Ο κόσμος πεθαίνει απλώς επειδή διαδηλώνει και πολλοί. Και προφανώς υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε με κανένα τρόπο. Και το τελευταίο είναι η κράτηση, η σύλληψη της Αμάγια Εύα Κόπενς που θα έχετε ακούσει ποια είναι που το Σεπτέμβριο ε, συνελήφθη και ε, κρατείται επειδή διαμαρτυρήθηκε κατά του καθεστώτος του Ντανιέλ Ορτέγα. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταστολή και τον εκφοβισμό των διαδηλωτών με αποτέλεσμα αυτό το τελείως απαράδεκτο που συνέβη. Επίσης θα πρέπει να απευθύνουμε πολύ ε, αυστηρή έκκληση ε, και πάρα πολύ έντονη προς τις αρχές της Νικαράγουας να σταματήσουν κάθε είδους βία κατά των διαδηλωτών. Τι κάνουν οι άνθρωποι, ασκούν ένα βασικό δικαίωμα εδώ στο Κοινοβούλιο δεν το αμφισβητεί κανεί την ελευθερία της έκφρασης. Και του συνεταιρίζεστε και του συνέρχεστε, αν είναι δυνατόν. Εδώ θα πρέπει γρήγορα να προβληματιστούμε γιατί έχει αλλάξει αυτή η τακτική και να το διερευνήσουμε κιόλας για το τι συνέβη πραγματικά. Βεβαίως να συνεχίσει ο εθνικός διάλογος με ειλικρίνεια, ανοιχτό. Όταν μιλάμε για ενότητα και συμφιλίωση, αυτά ακούγονται ηρωνικά καμιά φορά. Αλλά εσεί κύριε Πρέσβη, είπατε κάτι με το οποίο μπορώ να συμφωνήσω εν μέρη. Δεν νοείται ατιμορρησία για του ε, εγκληματίε. Συμφωνώ. Αλλά ούτε για εκείνου που δεν σέβονται τους νόμους, τα δικαιώματα και τι ελευθερίε. Ούτε για αυτού ατιμορρησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σημειώνω κάτι που είπατε. Είπατε ότι καλείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελειώνω, να βοηθήσει την Νικαράγουα. Βεβαίω, θέλει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Νικαράγουα. Αλλά να αφήσει και η Νικαράγουα να τη βοηθήσουν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να βοηθήσει. Γι' αυτό σήμερα το Κοινοβούλιο ενέκρινε ad hoc αντιπροσωπεία στην Νικαράγουα. Και ακολουθώ και τα λόγια σας. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα βοηθήσετε έτσι ώστε η δική μας αντιπροσωπεία που σήμερα εγκρίθηκε να είναι μια αντιπροσωπεία που να μπορούμε να τη βοηθήσουμε τη χώρα. Αλλά για να τη βοηθήσουμε θα πρέπει να έχουμε απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Να δούμε όποιον θέλουμε, να συναντηθούμε με όποιον θέλουμε και όπως πολύ καλά είπατε να βοηθήσουμε τη χώρα. Εκεί πάντα θα μας βρείτε σύμφωνος. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς κύριε συνάδελφε θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Πρέσβη και στην κυρία Φέλτα αν έχουν κάποιες τελικές παρατηρήσεις να κάνουν. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Πρέσβη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι η κυβέρνηση της Νικαράγουας έχει γνήσιο και αυθεντικό ε, ενδιαφέρον να προχωρήσω. Θα αφήσω στην πρόεδρο αυτό το έγγραφο για να είναι στη διάθεση της αντιπροσωπείας σας. Είναι η έκθεση της ε, ε, Επιτροπής Αλήθειας και Δικαιοσύνης για τα διάφορα αριθμητικά στοιχεία. 300-400 νεκροί ακούστηκαν. Σύμφωνα με τις ανακρίσεις και τις έρευνες που έγιναν από την αστυνομία και την εισαγγελία, έχουν προσθέσει εδώ τα τροχέα, τα θύματα από τροχέα, από επιθέσεις, από το κοινό έγκλημα εκείνη την περίοδο. Αυτά θα τα λύσει η ιστορία. Εδώ έχετε λεπτομέρειες και είναι στη διάθεσή σας κυρία Πρόεδρε και το μέλλον της αντιπροσωπείας. Βεβαίως, δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν και κρατούνται. Είναι αυτοί που κάνανε αυτά τα πράγματα. Καταστροφές, από αυτά που σας δείχνω. Δημόσιας περιουσίας. Έχετε εδώ φωτογραφίες παρακαλώ, τις οποίες σας παραδίδω και αυτές. Εδώ, κοιτάξτε. Και αυτό είναι ένα μόνο τμήμα των καταστροφών. Κάποιοι άλλοι που συνελήφθησαν, τι έκαναν. Απλοφορούσαν. Ορίστε, εδώ. Να, έτσι, αυτή είναι. Βεβαίως χρειάζεται δουλειά, με σοβαρότητα για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο δρόμο της ειρήνης και της σταθερότητας. Σας ευχαριστώ την αντιπροσωπεία σας για το ενδιαφέρον και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ενδιαφέρον. Σημειώνω τις παρατηρήσεις που κάνατε. Θα το διαβιβάσω, όπως πάντα, ότι ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξελίξεις και στην Ικαραγώα και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως μπορέσαμε και στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, κύριε Μάτα, έχετε το λόγο. Sí. Ναι, πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Δυστυχώς εγώ να δείτε φωτογραφίες που θα ήθελα να σας δείξω. Αλλά πολλές, ε, πολλοί από αυτούς των φωτογραφιών είναι ή δολοφονημένοι ή φυλακισμένοι. Τι να σας δείξω. Είναι θλιβερό να συζητάμε για νεκρούς. Έστω και ένας να είναι επειδή έχει ζητήσει την ελευθερία. Μην λέμε τώρα για τροχέα και τέτοια. Αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Έχετε κάποια παρατήρηση κυρία No, unless there's a... Όχι. Εκτό και αν υπάρχει κάποια ερώτηση για μένα. Ευχαριστώ. Νομίζω πω δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, οπότε σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και κύριε Άφερτ. Και συνάδελφε, πάμε στο πέμπτο σημείο τη ε, σημερινή μα ημερήσια διάταξη που αφορά την επίσκεψη αντιπροσωπεία μα στην Κεντρική Αμερική κατά την 44η εβδομάδα του χρόνου, δηλαδή από 29 μέχρι Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου. Όπως γνωρίζετε, στην διάσκεψη των Προέδρων της 31ης Μαΐου του 2018 εξουσιοδοτήθηκε η προσωπία μας να επισκεφθεί την Κούβα αυτή την εβδομάδα που ανέφερα προηγουμένως. Στο διάστημα αυτό ζήτησα επανειλημμένα προσωπικά αλλά και μέσω της Γραμματείας επίσημη επιβεβαίωση από την κουβανική πλευρά για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της συγκεκριμένης αποστολής. Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αβάνα, ο κύριος Ναβάρο, ενημέρωσε τη γραμματεία της αντιπροσωπείας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας ζήτησε να αναβληθεί η επίσκεψη για μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς η Κουβανική Εθνική Συνέλευση δεν μπορεί να δεχθεί την αντιπροσωπεία μας στις προτινόμενες ημερομηνίες. Ο κύριος λόγος που προβλήθηκε για την αναβολή της επίσκεψης ήταν η δημόσια διαβούλευση για το νέο σχέδιο συντάγματος της Κούβας, η οποία λήγει στις 15 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Σας υπενθυμίζω ότι κατά τις Τις προηγούμενες συνεδριάσεις αντιπροσωπείας είχε προταθεί από τα μέλη της αντιπροσωπείας ότι σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης επίσκεψης στην Κούβα, ελπίζω ότι θα το θυμόσαστε, θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στην Ικαράγουα και στην Γουατεμάλα. Να σας θυμίσω επίσης ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της αντιπροσωπείας, ο πρόεδρος της Eurolat, ο κύριος Χαουρέγγι, επανέλαβε το αίτημα να πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στην Ικαράγουα. Με βάση τα αιτήματα των μελών της αντιπροσωπείας, επανέλαβα κατά την προηγούμενη διάσκεψη ότι αν δεν πραγματοποιηθεί η αποστολή στην Κούβα, θα ζητηθεί να γίνει στην Ικαράγουα και τη Γουατεμάλα κατά την 44η εβδομάδα του Οκτωβρίου πρόταση που έγινε αποδεκτή από τα μέλη. Λόγω των ασφικτικών προθεσμιών, πήρα την πρωτοβουλία και απέστειλα επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων, με την οποία την ενημέρωνα ότι η Επιτροπή μα σκοπεύει να ζητήσει αποστολή στι δύο χώρε που ανέφερα. Δυστυχώ, η επόμενη διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία θα αποφασιστεί η πρόταση τη ΔΕΚΑΜ, θα πραγματοποιηθεί στι 18 Οκτωβρίου του 2018. Τα χρονικά περιθώρια λοιπόν είναι ασφικτικά και θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα αν θέλουμε να γίνει επίσκεψη στις, ε, μα στι μας στις που αναφέρθηκα προηγουμένως. Θα ήθελα, <laughs> κύριε συνάδελφε, να ζητήσω να τοποθετείτε αν έχετε κάποιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα κάποια θέση. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριο Σμάτο. Καταρχάς, λυπάμαι αλλά δεν με εκπλήσει. Είναι η πέμπτη φορά που μας αρνούνται τη δυνατότητα να πάμε στην Κούβα. Και καθυστερεί αυτό, καθυστερεί, καθυστερεί. Εμείς δεν καθυστερήσαμε την έγκριση του διαλόγου. Είναι περίεργη αυτή η κατάσταση. Μπορούν οι πάντες να πάνε στην Κούβα εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι περίεργο αυτό είπαμε ότι θέλουμε να πάμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να επισκεφθούμε την Κούβα όπως θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, σας το έχω ξαναπεί και τις άλλες φορές που είπατε να πάμε στην Κούβα. Να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις, γιατί δεν μας αφήνουν να πάμε στην Κούβα. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά ξέραμε ότι δεν μας αφήνουν να πάμε. Ε, δεν έχουμε την ελευθερία μας. Ε, θα υπάρξει άλλη επίσκεψη. Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να κάνουμε αυτές τις επισκέψεις. Το να πάμε σε δύο χώρες είδαμε από την πείρα μας ότι είναι πολύ μικρός ο χρόνος και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού πηγαίνει ad hoc αντιπροσωπεία στην Νικαράγουα, μήπως η αντιπροσωπεία μας να πάει μόνο στη Γουατεμάλα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με χαρά να πάω και στην Νικαράγουα όσες φορές χρειαστεί και πάντα ε, με σύνθημα την απόλυτη ελευθερία να βρούμε και να δούμε όποιον θέλουμε και όποιον θεωρούμε εμείς χρήσιμο και σκόπιμο. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, δεν έχω καμία αντίρρηση να δεχθώ την οποιαδήποτε πρόταση. Οφείλω όμω να ομολογήσω, οφείλω να πω και να επισημάνω ότι είχαμε πει ότι πριν γίνει αυτή η ad hoc αποστολή, ε, πριν γίνει αυτή η ad hoc αποστολή, έπρεπε να περιμένουμε την απάντηση της, uh, Κούβας και θα αποφασίζαμε αμέσως μετά να πάμε σε Νικαράγουα και Ελσαλβαδόρ. Ε, δυστυχώς, κάποιοι τρέχουν τα θέματα πολύ διαφορετικά από ό,τι τα αποφασίσαμε μέσα αυτήν την αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι είναι στη δική μας, παραμένει στη, δική μας επιλογή το ποια χώρα θα επιλέξουμε να πάμε, γιατί η, η, Επιτροπή μας θα πρέπει να κάνει μια επίσκεψη σε αυτές τις χώρες. Νομίζω θα περιμένω από εσά από όλα τα μέλη μάλλον της, ε, Επιτροπής την, ε, την πρόταση που θα μπορούσα να μου κάνω όσον αφορά την χώρα της επίσκεψης θα έπρεπε να, να επιλέξουμε. Αυτό. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. <laughs> Ε, Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. <laughs> Η ομάδα μας θεωρεί το εξής. Εμείς πήγαμε στην Κούβα σε άλλες αποστολές και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει τώρα άνοιγμα από την Κούβα και είναι ένα κράτος κυριαρχό σε πλήρη διαδικασία νομοθετική με την Λαϊκή Εθνική Συνέλευση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ε, είναι θέμα χρονικό. Ε, γίνεται λόγος για την ΤΕΚΑΜ, για τις προτάσεις και εμείς Πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη στη Γουατεμάλα αυτή τη στιγμή και χρειάζεται να πάμε για διάφορους λόγους. Πρώτον, υπάρχουν περιπτώσεις δολοφονιών αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την περασμένη εβδομάδα η κυρία Χουάνα Ραμύρες, ε, ακτιβίστρια και υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρο, Φιλολίτα Τσάβεθ. Αυτή τη στιγμή αγνοείται η τύχη της δεν ξέρουμε που βρίσκεται, μπορεί να γυρίσει στη Γουατεμάλα. Χρειάζεται ε, σεβασμός και δεν είναι μόνο ότι ήταν υποψήφιο για το βραβείο Ζαχάροφ, αλλά να παρατηρήσουμε τι γίνεται στην κατάσταση. Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας αποφάσισε να μην ανανεώσει ε, την ε, εντολή της Διεθνούς Επιτροπής ε, κατά της ατιμορρησίας της Γοτεμάλας. Και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τα ξέρει αυτά και αμφισβητεί την απόφαση αυτή της Γοτεμάλας να μην ανανεωθεί εντολή της ε, λόγω επιτροπής. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο οργανισμός αυτός που δημιουργήθηκε ακριβώς μετά από αίτημα της κυβέρνησης της Γοτεμάλας ε, βοήθησε για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας και της διαφθοράς. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσει το έργο της και να μεταβεί εκεί η αντιπροσωπεία για να επαναληφθούν οι εργασίες της Επιτροπής αυτής. Διεθνής Επιτροπή, επαναλαμβάνω, κατά της ατιμορρησίας. Έχουμε υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ και ε, Άλλε γυναίκες, πρέπει να πάμε στη Γουατεμάλα. Ευχαριστώ. κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριο Μάτο, να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέει η κυρία Μιράντα εμείς, σε ποιον αναφέρεται. Η άκρα αριστερά μπορεί να πάει στην Κούβα όποτε θέλει, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14-15 χρόνια δεν μπορεί να πάει στην Κούβα. Εγώ μιλάω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν λέω εμεί. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα. Εγώ και έχω προτείνει και Γουατεμάλα εδώ και καιρό. Το λέει και στα πρακτικά. Δεν ξέρω από πότε προτείνω Γουατεμάλα. Ε, εν πάση περιπτώσει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία να πάμε στη Γουατεμάλα. Θαυμάσια πρόεδρε, αν το θεωρείτε σκόπιμο. Κύριε συνάδελφε, προσωπικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ακρά αριστερά. Στη, στην ε, Κούβα πάντως έκανα επίσκεψη και πραγματικά ήταν ε, πολύ εντυπωσιακό και πολύ ενημερωτικό για μένα. Ε, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι και, και στην κυρία συνάδελφα αλλά και στην Επιτροπή και όπω αναφέρθηκα στην αρχή τη κουβέντα μα, στη Γουατεμάλα έχουμε ξαναπάει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αφού υπάρχει πρόταση να επισκεφθούμε τη Γουατεμάλα. Είναι μια χώρα, α πούμε, ότι έχει κλειδώσει. Από εκεί και πέρα η γραμματεία με τι αντιπροσωπείε θα συζητήσει για να βρούμε και τη δεύτερη χώρα που θα μπορέσουμε να κάνουμε το συνδυασμό αυτό για να ολοκληρωθεί η επίσκεψή μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν θέλετε, γιατί από ό,τι φαίνεται είμαστε δύο βουλευτές εδώ και εσείς Πρόεδρε να αφήσουμε 24 ώρες για να το δουν οι πολιτικές ομάδες και να κάνουν μια πρόταση αν θέλετε. Ε, εντάξει, πάντως θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτές τις ε, επισκέψεις η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη να κάνει μια επιστολή προς τους Κουβανούς τουλάχιστον να εκφράζει την ε, ε λύπη της δεν ξέρω με ποια σκληρότητα θα το γράψει. Για μένα θα ήταν πολύ πιο βαριά η επιστολή από ό,τι θα τη γράψει η ίδια. Μετά από 15 χρόνια ε, έχουμε λαχταρίσει να πάμε στην Κούβα από ό,τι λένε είναι όλο και πιο ελεύθερη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τα ονόματα, για τους αριθμούς μάλλον, η ομάδα μας θα μπορούσε να σας δώσει 120 ονόματα πολιτικών ε, ε, κρατουμένων, κουβανών, που είναι στις κουβανικές φυλακές και κρατούνται παράνομα. 120, μόνο και μόνο επειδή έχουν δημοκρατικά φρονήματα. Κύριε Μιράντα, ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι για τα όσα είπε ο κύριος Μάτο για το ποιοι είμαστε εμείς όταν λέω εμείς. Εμείς είμαστε αριστεροί. Τώρα ακροαριστεροί δεν ξέρω. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς κρατήστε τους, γιατί από πλευρά δημοκρατίας δεν έχουμε μαθήματα να παίρνουμε. Είδαμε πώς ψηφίσατε για την Ουγγαρία για το άρθρο 7. Μην χάνετε και χαρακτηρισμούς τώρα. Κύριε να το κλείσουμε γιατί πολύ ωραίο. Δεν θα μπω σε αυτό το θέμα γιατί η κυρία Μιράντα προφανώς ε, αυτό χαρακτηρίζεται. Και ε, είναι περίεργο. Γιατί τέτοια λαχτάρα για να υπερασπίζετε την Κούβα και με τέτοια λαχτάρα και μανία να επιτίθεται σε άλλες χώρες. Εν πάση εμένα δεν με νοιάζει. Να πάμε όπου θέλετε. Αν θέλω, εγώ θέλω να πάω στην Κούβα, αλλά να με αφήσουν να πάω. Δεν είναι, δεν είναι περίεργο πράγμα. Να με αφήσουν να πάω στην Κούβα που δεν με αφήνουν. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο αυτό ζητάω, τίποτα άλλο. Και τα δεξιά-αριστερά δεν με νοιάζει. Αφήστε το Κοινοβούλιο να πάει στην Κούβα που νομίζω ότι είναι δημοκρατικό. Τι ζητάμε πια. Δεν ξέρω, τον ουρανό μετάστρα. άστρα ζητάμε. Λοιπόν, προσωπικά πιστεύω ότι και στην Κούβα θα πάμε όταν θα έρθει η ώρα και όταν θα έχουν τελειώσει τι διαδικασίε που οι ίδιοι έχουν βάλει και όσον αφορά την ανα το Σύνταγμά του. Ε, αυτό που θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, να κλείσουμε τη συνεδρία, η οποία ήταν σε καλό κλίμα, να μην το χαλάσουμε τώρα στο τέλο. Και ότι η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπεία μα θα πραγματοποιηθεί την 5η στι 11 Οκτωβρίου του 2018 στι Βρυξέλλε. Να σα ευχαριστήσω όλου, και εσά κύριε Γουάτζη, ε, για την παρουσία σας, για τις, παρεμβάσει για τις παρεμβάσεις σας και για το όσα υπόθηκαν. Ευχαριστήσω και τους διερμηνούς για την ε, υπέρβαση που κάνανε στον χρόνο και για την βοήθεια που μας δώσαν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.